Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω θερμά. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουμε τις ε, δηλώσεις του Συμβουλίου για την παρουσίαση του προγράμματος ε, της Τσεχικής Προεδρίας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Μίρεκ Τοπολάνεκ, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Σας καλωσορίζουμε θερμά, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τοπολάνεκ. Επίσης, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά και τον κύριο Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όλοι μας ε, γνωρίζουμε ότι η Προεδρία είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργό κύριος ε, Τοπολάνεγκ ε, και πνευματικά αλλά και συναισθηματικά το εκλαμβάνει την Προεδρία ως πρόκληση ε, διότι έχει ζήσει τα χρόνια του κομμουνισμού και τώρα ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργεί πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη Σλοβενία αυτή είναι η δεύτερη Προεδρία μιας χώρας η οποία προσεχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Και φαντάζομαι εξ όλων μπορώ να πω ότι η τσεχική Προεδρία ε, χέρι της αμέριστης υποστήριξής μας και επιθυμούμε όλοι διακαώς σε τόσο δύσκολες εποχές η Τσεχική Προεδρία να στεφθεί από επιτυχία. Μετά από αυτά θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τοπολάνεκ να απευθύνετε το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε θερμά στο χώρο αυτό. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.